και στην οικονομική, κοινωνική και οικονομική ζωή και στην οικογένεια με τις ε, καλύτερες ε, επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φιγερέδο. Ολοκληρώσαμε αυτή τη συζήτηση. Ήταν προνόμιο να είμαι πρόεδρος σε αυτή τη συζήτηση. Όχι μόνο για τον αριθμό των ατόμων και συναδέλφων που ήταν παρόντες και παρούσες, αλλά επειδή ήταν υποδειγματικός ο ρόλος και η συμμετοχή. Η πλειοψηφία των ε, συμμετεχόντων ήταν παρόντες εδώ και παρούσες από την έναρξη της συζήτησης μέχρι το τέλος Απλά αυτό είναι ασυνήθιστο, δεν γίνεται κάθε φορά. Όλοι ήταν παρόντες και άκουγαν τις σημαντικές παρεμβάσεις των άλλων. Δεν ήρθαν μόνο να κάνουν την παρέμβασή τους και να φύγουν και να ε, περάσουν μετά από την, είσοδο, την έξοδο και να φύγουν, αλλά έμειναν. Ακούσαν τους συναδέλφους που παρενέβαιναν, συμμετείχαν όπως αναμένεται από πραγματικούς κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, αυθεντικούς ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ όλους σας λοιπόν, γυναίκες και άντρε. Η ψήφιση αυτών των θεμάτων θεμάτων που συζητήσαμε απόψε θα γίνει αύριο το μεσημέρι. <clears throat> Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλες και όλους. Το ακόλουθο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση που υποβάλλει η κυρία Εκ για το κοινό πρόγραμμα, πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης για τη Βαλτική θάλασσα. Θα λάβει τώρα τον λόγο υπό την ιδιότητα ε, εισηγήτριας η κυρία Εκ. Τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προσέξτε. Ισπανική Προεδρία φυσικά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η Βατική θάλασσα χρόνια πριν από μια καθαρή θάλασσα που ήταν πέρασε σε μια θάλασσα, θαλάσσια περιοχή που έχει πλέον μολυνθεί ε, και βρίσκεται σε δινή κατάσταση. Ε, δηλητηριώδεις ουσίες, απόβλητα, η μόλυνση έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση που είναι ολέθρια στη Βαλτική παρόλες τις πρόοδους ε, που σημειώθηκαν στη δεκαετία του 90 έχουμε περιεκτικότητα αζότου που έχει περιοριστεί ακόμα περισσότερο. Υπάρχει υπερβολική ε, λιπαντές και λιπάσματα ε, εκβάλλουν στην Βαλτική θάλασσα και έχουμε περιεχόμενο ε, που παρότι όσον αφορά τον υδράργυρο ε, έχει μειωθεί, άλλες δηλητηριώδεις ουσίες έχουν αυξηθεί. Αυτή η κατάσταση στη Βαλτική θάλασσα είναι χαρακτηριστική. Όταν πάει κανείς ε, με τη βάρκα του ε, και βλέπει ένα μέτρο ολόκληρο ε, πυκνής επιφάνειας με, διάφορα, με διάφορες άλγες και φύκια και προσπαθούν κάποιοι να περάσουν από αυτή την θα έλεγε κανείς συμπαγή μάζα και βλέπουν ότι και τα ψάρια δεν μπορούν να αντέξουν και ε, ψοφάνε. Είναι μια κατάσταση πραγματικά ολέθρια. Πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση στη Βαλτική θάλασσα. Τα οικοσυστήματα στη Βαλτική είναι πολύ σύνθετα και περίπλοκα. Για να τα κατανοήσουμε χρειάζεται διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ε, κοινοτήτων και ομάδων ερευνητών. Υπάρχει αυτή η έρευνα σήμερα, αλλά δεν επαρκεί δυστυχώ. Δεν υπάρχει επαρκή συνεργασία και συντονισμό. Και για να αλλάξουν όλα αυτά, έχουμε τη σημερινή πρόταση που υποβάλλεται. Ε, και προσπαθούμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό πρόγραμμα έρευνας των ε, ομόρων κρατών ε, της, στη Βαλτική συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας σε αυτό το πλαίσιο. Το bonus είναι ένα στρατηγικό πλαίσιο ε, που συμπεριλαμβάνονται 500 ερευνητές των ομόρων κρατών ε, της Βαλτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όμορα κράτη σχεδόν ένα δισεκατομμύριο κορώνες, σουηδικές κορώνες ε, θα επενδύσουν. Έχουμε 85 εκατομμύρια οίκων γύρω από την Βαλτική και η οικονομία όλων αυτών των χωρών εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την ίδια τη Βαλτική. Αν υπάρχουν απόβλητα τα οποία καταλήγουν στη Βαλτική αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις για όλους. Η έρευνα σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ κατακαιρματισμένη. Είναι ακόμα πολύ ε, θα έλεγα ε, τμηματική και εμβαλωματική. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τον εθνικό χαρακτήρα της έρευνας ενώ υπάρχει ανάγκη για ένα υπερεθνικό ερευνητικό πλαίσιο θα πρέπει εδώ τα κράτη τα οποία θα συμμετέχουν να μπορέσουν για πρώτη φορά να καταλήξουν σε ένα κοινό στρατηγικό πρόγραμμα με σαφή ε, κέντρα βάρους. Ευχαριστώ όλους ε, που συνεργάστηκαν και σε σχέση με τους συναδέλφους αλλά και την Ισπανική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε όλοι αυτοί οι στόχοι να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν και να λειτουργήσουν σωστά. Πρόκειται για θέμα αηφορίας, ε, για τη διαμόρφωση των πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η αηφορία. Η Βαλτική θάλασσα είναι πολύ σημαντική. Έχει αποφασιστικό ρόλο για όλες αυτές τις χώρες που είναι όμορες χώρες. Υπάρχει και μακρά παράδοση θα έλεγα σε σχέση με πολιτισμικά θέματα. Ούτως ή άλλως θέλουμε να διατηρηθεί αυτή η κληρονομιά στα παιδιά μας και το πόνους θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο. Εξ ονόματος της Επιτροπής λέγει ο Πρόεδρος ε, η κυρία Γκέγκεν τον λόγο, που πάλι την καλωσορίζουμε, γιατί όσο με αφορά δεν είχα ευκαιρία να προεδρεύω σε μια συζήτηση όπου να παρεμβαίνει η ίδια. Καλώς ήρθατε και έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ε, Vice Αντιπρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο Ευρωκοινοβούλιο ε, και στην εισηγήτρια κυρία Έκα που υποστήριξε την πρόταση της ε, κοινότητας για το κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξη στη Βαλτική θάλασσα Μπόνους. Έχουμε επικοδομητική υποστήριξη και επίσης η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε το πρόγραμμα Bonus. Νέα κράτη παράκτια της Βαλτικής έχουν σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της Βαλτικής και των προβλημάτων που ανέφερε τόσο εύγολα η συγγήτρια. Αυτό ε, απειλεί την ικανότητα των χωρών της Βαλτικής να παρέχουν τις υπηρεσίες από τις οποίες όλες εξαρτώμεθα. Η επιστήμη παίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα της έρευνας και του περιβάλλοντας. Όμως ο κατατεμαχισμός και η έλλειψη συντονισμού και συνεκτικότητας και συνοχής έχει υπονομεύσει την αποδοτικότητα. Αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή της Βαλτικής. Είναι σαφές ότι καμία χώρα μόνη δεν μπορεί να επιτύχει για να επιλύσει τα περίπλοκα περιβαλλοντικά θέματα της περιοχή Για να ανταπιστούν αυτά τα προβλήματα της Βαλτικής είναι πήγον τώρα να αναπτύξουμε ε, μια στρατηγική ολοκληρωμένη ε, που να επιτρέπει συνέργειες διασυνοριακές, ε, μοίρασμα των πόρων, καταμερισμό του φόρτου εργασίας για να υπάρχει ένας διατηρήσιμο μέλλον για την Βαλτική. Η πρωτοβουλία Μπόνους και οι, οι ε, πρωτοβουλίες μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής θα επιτρέψουν να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές με τρόπο συντονισμένο και επικοδομητικό. Είχαμε μια θεσμική συμφωνία για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας Μπόνους 27 Απριλίου. Τούτων λεχθέντων θα ήθελα να τονίσω την λύπη μου και την έλλειψη συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών για την θέσπιση ενός κοινού μοντέλου όπως είχε αρχικά λεχθεί στην αρχική πρόταση Κομισιό χωρίς να έχουμε μια κοινή ευκολία χρηματοδότησης. Οι προτάσεις συνοριακές έρευνες που βασίζονται στην αριστεία, την επιστημονική, την ποιότητα του κονσόρτσιουμ δεν μπορούν να εξασφαλιστούν. Δεν επιτρέπεται η πλήρης υλοποίηση και αξιοποίηση του ωφέλους μιας διασυνοριακής συνεργασίας. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι οι συνέπειες της απόφασης δεν πρέπει να θεωρηθούν προηγούμενα για μελλοντικές αποφάσεις. Τα κράτη-μέλη πρέπει να δεσμευθούν για διασυνοριακή χρηματοδότηση και συνεργασία πρώτου υπάρξει νέα πρωτοβουλία βάσει του άρθρου 185 της Συνθήκης Λίσσα Σχετικά με την τρέχουσα πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πεπισμένη ότι το πρόγραμμα Bonus θα μπορέσει να βελτιστοποιήσει τα προγράμματα περιβαλλοντικά στον τομέα της Βελτικής, να προωθήσει τις ικανότητες οι επιστημονικές στις περιοχές, να, ε, να προωθήσει την κινητικότητα των ερευνητών, τις συνέργειες και τις προσπάθειες για να υπάρξει ένα διατηρήσιμο μέλλον για την Βαλτική. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε εξ ονόματο τη Επιτροπής Περιβάλλοντος. Για ένα λεπτό η κυρία Ρόσπαχ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μπόνους και 169. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα, για ένα σημαντικό εγχείρημα. Πρόκειται για τη συνεργασία σε σχέση με περιβαλλοντικά προβλήματα και την υπέρβασή του στην Βαλτική. Αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις όμορες χώρες ε, της Βαλτικής και σε σχέση με την ε, κατάθεση αποβλήτων στην Βαλτική θάλασσα που είναι μία από τις πιο επιβαρημένες θάλασσες παγκόσμια. Αυτό το πρόγραμμα έχει ένα πολύ μεγάλο στόχο όλα αυτά τα προβλήματα στη Βαλτική να τα απαριθμίσει, να τα διερευνήσει και να τα ε, αντιμετωπίσει. Υπάρχουν ε, χαρτοβιομηχανίες, οι τα αποθέματα ηχθείων ε, αποβιώνουν, υπάρχουν μεγάλη αγωγή φυσικού αερίου που διέρχονται, διασχίζουν τη Βαλτική. Για όλους αυτούς τους λόγους χρειαζόμαστε το πρόγραμμα Bonus, αλλά δεν πρέπει να απομείνει μόνο του, απομονωμένο. Πρέπει από τα κράτη-μέλη να υποστηριχθεί με τον δέοντα τρόπο για να είμαστε αποτελεσματικοί. Χρηματοδοτικά φυσικά, όχι μόνο με την πολιτική βούληση. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι. Περνάμε τώρα στον γύρο των παρεμβάσεων εξ ονόματος των ομάδων. Πρώτα απ' όλα εξ ονόματος του ΕΛΚ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Φανίστερ Ρόι. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τα ειδικά προβλήματα της Βαλτικής θάλασσας απαιτούν μια προσέγγιση ιδιαίτερη και στοχοποιημένη. Νομίζω ότι μπορούμε τώρα να κλείσουμε με όσα είπαμε, με τα λόγια και να στρωθούμε στη δουλειά. Αυτό που είπε και η Επίτροπος, θέλουμε ε, μια συζήτηση σε βάθος για να δούμε τον απολογισμό και μετά να δούμε τα κριτήρια αριστείας, τα, τους διάφορους τομείς που να δούμε το θέμα πολυκλαδικά. Μετά γίναμε πιο ρεαλιστές, είπαμε ότι το κάθε χώρα μπορεί να διαλέξει από τα προγράμματα των πανεπιστημίων. Δεν έχουμε καμιά αντίρρηση, αλλά πρέπει όσο να είναι να εξελιχθούμε, να γίνει όλα αυτά με τρόπο αποτελεσματικό και καλύτερα από το παρελθόν ούτως ώστε να αποτελέσει η προσπάθεια αυτή παράδειγμα για το τι θέλουμε για την στρατηγική 2020. Η Ευρώπη πληρώνει, τα κράτη-μέλη πληρώνουν, αλλά δεν θα πρόκειται μόνο για έρευνα, αλλά και μετά για την υλοποίηση, την εκτέλεση ούτω ώστε να αποκατασταθούν οι συνθήκες οι που επιθυμούμε. Δύο παρατηρήσεις. Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση στην Βαλτική μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες περιοχές και αναφέρομαι στο Δούναβι παραδείγματος χάρη και ρωτώ την Επίτροπο μήπως δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε την περιοχή αυτή. Σα ευχαριστούμε. Εξ ονόματο τη Σοσιαλιστική Ομάδα για δύο λεπτά θα λάβει τον λόγο ο κύριο ε, Γκέμπερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, το σχέδιο πρότασης που αφορά την απόφαση για την ε, εξυγίανση της Βαλτικής ε, εμπεριέχει ένα σημαντικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού. Χωρίς αυτό θα είχαμε μόνο μια απλή επέκταση έρευνας. Ε, χρειάζεται ένα πρόγραμμα δράσης με καλύτερη στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη Βαλτική θάλασσα, αλλά επίσης ε, και τις λεκάνες, τις ε, όμορες λεκάνες. Η επιλογή των ε, ερευνητών ε, και οι ερευνητικές δράσεις ξεπερνούν την, τις δοκιμασίες σε εργαστήρια. Έχουμε εδώ και την δικαιοδοσία των όμορων χωρών. Όλα αυτά θα πρέπει να αναφέρονται στην επιλογή από πλευρά επαϊόντων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανεξαρτήτων επαϊόντων. Όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τα εξή στοιχεία. Πρώτον, δυναμικό έρευνας στα κράτη διακυμαίνεται φυσικά και σε σχέση με αυτό βαίνει εκ παραλίλου με τις ε, δυνατότητες ε, ερευνητικές δραστηριότητες ε, της κάθε χώρας. Γι' αυτό έχουμε και ένα συγκεκριμένο ποσοστό στη συμμετοχή έρευνας από τις χώρες. Δεύτερον, όχι μόνο είναι νομικά απαράδεκτη μια τέτοια επιπτώση, θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και στα ερευνητικά σχέδια. Τρίτον, η στρατηγική αυτή ευδοκίμηση απαιτεί χρόνο. Θα πρέπει να γίνει καλύτερη χρήση και όσον αφορά τις δυνατότητες που αναφέρονται στην πρόταση. Πρώτον θα πρέπει να υπάρξουν προτεραιότητες ερευνητικές ε, για τη Βαλτική και μόνο τότε όταν θα έχουν καθοριστεί αυτές οι προτεραιότητες να εξειδικευτούν οι δράσεις ε, με μέσα ερευνητικά. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκέρεκ, εξ ονόματος ε, των Πρασίνων Χασί. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τους την εισηγήτρια κυρία Λένα Έκε για την εξαιρετική δουλειά που επετέλεσε. Αυτό το πρόγραμμα, το ερευνητικό πρόγραμμα Bonus, το οποίο θα υποστηριχθεί και πρέπει να υποστηριχθεί είναι μια απόρρια της στρατηγικής για τη Βαλτική από Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο προόδου η Βαλτική θάλασσα ε, έγινε, η Βαλτική έγινε μια ε, θάλασσα της ε, κοινότητας με την διεύρυνση. Όμως όπως διαπιστώθηκε έχει, έχουν γίνει αρκετές ερευνητικές δράσεις στη Βαλτική αλλά υπάρχει πολύ μικρή συνιστόσα συντονισμένων δράσεων εκεί, ώστε να είμαστε πιο ευφυείς και πιο δημιουργικοί σε σχέση με τον συντονισμό της έρευνας. Ελπίζω ότι με τη συντονισμένη έρευνα δύο πράγματα θα μπορέσουμε να δούμε και να διερευνήσουμε. Πρώτον, για ποιους λόγους είναι ανησυχητική η οικολογική κατάσταση της Βαλτικής, που είναι μία από τις πιο μολυσμένες θάλασσες παγκόσμια. Έχουμε τον ευρύτερο πυθμένα που είναι ο ευρύτερος πυθμένας χωρίς ε, άζωτο και βλέπουμε ότι είναι ο πιο μολυσμένος πυθμένας ε, θάλασσας ε, Επίσης, εκείνο το οποίο εμείς πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι εμείς είμαστε ένοχοι για αυτή την κατάσταση. Φταίμε εμείς. Ο ευτροφισμός είναι μια άλλη περίπτωση που συναντάται στη Βαλτική η μεγαλύτερη πηγή, το μεγαλύτερο αίτιο για τα φωσφορούχα είναι τα λιπάσματα τα οποία εκβάλλουν, εκβάλλονται στην ε, Βαλτική μαζί με άλλα απόβλητα. Ελπίζω ότι με ένα ε, συντονισμένο πλαίσιο έρευνας θα κατανοήσουμε καλύτερα αυτά τα φαινόμενα θα τα ερευνήσουμε και θα βρούμε καλύτερες μεθόδους, ευφιέστερες μεθόδους για όλους αυτούς τους κλάδους και τομείς. Έχω υπόψη σφαιρικότερα τη γεωργία. Τα λιπάσματα τα οποία καταλήγουν στους ποταμούς και μετά που εκβάλλουν στη θάλασσα είναι σίγουρα μια διασπάθηση ε, για τους ε, γεωργούς. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι η έρευνα δεν επαρκεί αφέ αυτής. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η διάσωση της Βαλτικής απαιτεί αλλαγή στις πολιτικές μας, εκβάθρων αλλαγές, κυρίως στη γεωργία αλλά και σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων μας, στις πολιτικές μας. Ελπίζω λοιπόν ότι εμείς θα καταφέρουμε τη Βαλτική να την κάνουμε, σε, να οδηγηθεί σε μια επιτυχία ώστε και οι, επόμενοι, οι επόμενες γενναίες να μπορέσουν να μάθουν. Περνάμε τώρα στις παρεμβάσεις ατομικά από τους Ευρωβουλευτές. Για 1,5 λεπτό η κυρία Καρβάλιο πρώτη παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, εκφράζω την ικανοποίησή μου και συγχαίρω για το πρόγραμμα Bonus για το συντονισμό των εθνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο περιβάλλον και στη διαχείριση των ε, θαλάσσιων πόρων στη Βαλτική. Το πρόγραμμα Bonus ε, είναι ένα υπόδειγμα και αποτελεί κίνητρο και για άλλες ε, μορφές περιφερειακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. <clears throat> Η ε, περιοχή της Βαλτικής και άλλες ε, περιφέρειες όπως για παράδειγμα στην ε, νοτιοανατολική Ευρώπη και στην νοτιοδυτική Ευρώπη θα ε, ήταν υποφελής η διεύρυνση αυτής της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να μπορέσουμε την αηφόρο ανάπτυξη να τη βασίσουμε σε αυτές τις δράσεις των περιφερειών μας. Και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζοντας αυτή τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα για την ε, περιοχή αυτή της Ευρώπης ε, λαμβάνοντας υπόψη περιοχές ε, τομείς ιδιαίτερης σημασίας, τη θάλασσα, της την αηφόρο ανάπτυξη του Ατλαντικού άξονα της Ευρώπης ε, και των ε, θαλάσσιων παράκτιων περιοχών ε, των χωρών που βρίσκονται σε αυτή την νοτιοδυτική περιοχή της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε αυτό το γύρο. Έχουμε τέσσερις συναδέλφους στο Catch the Eye. Στο ένα λεπτό θα αφαιρώ το μικρόφωνο. Ο κύριος Λούχαν έχει πρώτο τον λόγο. Παρακαλώ. Domnule președinte, implicarea comunității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 ασχοληθεί περισσότερο με τη Βαλτική ε, θάλασσα, χρειάζεται κοινή κοινοτική δράση για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος με ενσωμάτωση όλων των πρωτοβουλειών σε ένα ενιαίο πρόγραμμα. Και αυτό για να εξασφαλίσουμε την αηφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ θετικό για την περιοχή της Βαλτικής, αλλά δεν θα πρέπει το πρόγραμμα να στοχεύσει μόνο την ε, περιοχή αυτή. Αυτή η μορφή περιφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές όπως στη Μεσόγειο και γιατί όχι και στον Δούναβι. Έτσι μόνο θα έχουμε μια ε, ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Μορκουνάιτε. Κύριε Πρόεδρε, η εφαρμογή του προγράμματος επιστημονικής έρευνας στη Βαλτική έχει αποκαλύψει την καταστροφική κατάσταση στην οποία ε, βρίσκεται η Βαλτική ε, θάλασσα. Και το πρόγραμμα αυτό ε, εφαρμόζεται όχι μόνο από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από άλλες χώρες. Η ε, τοξικότητα ε, σε ορισμένες περιοχές έχει αυξηθεί κατά εκατοντάδες φορές. Το πρόγραμμα Bonus θα συμβάλλει στην παρακολούθηση της Βαλτικής θάλασσας, ούτως ώστε η έρευνα να γίνεται με αποτελεσματικό και αντικειμενικό τρόπο. Και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί συμμετοχή επιστημόνων και από από ε, τις άλλες χώρες. Και επίσης ε, ε, χρειάζεται η κατάλληλη χρηματοδότηση ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και να αποφευθούν οι οικολογικές καταστροφές. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ τα προβλήματα θα μπορέσουν να επιληθούν με καλύτερο τρόπο αν οι ερευνητικέ δραστηριότητε των κρατών μελών ε, γίνονται με ε, κοινό και συντονισμένο τρόπο. Και γι' αυτό ε, είναι πολύ καλή η πρόταση για το bonus 169. είναι γεγονός ότι η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση του προγράμματος ώστε να κριθεί η αποτελεσματικότητά του και το κατά πόσο να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Τα αποτελέσματα αυτά θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος και έτσι οι επιχειρήσεις μπορούν να πληροφορηθούν ε, τα σχετικά ε, που χρειάζονται για να σχεδιάσουν τις ε, επενδύσεις τους. Ε, με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η προστιθέμενη αξία που θα έχει το πρόγραμμα αυτό για τις επιχειρήσεις, για την περιοχή, για το περιβάλλον, ιδίως στα πλαίσια της σημερινής κρίσης. Ο κύριος Σιτέσκι. Κύριε Πρόεδρε, ε, εγκρίνω 100% ε, το πρόγραμμα αυτό ε, για τη Βαλτική, το πόνους 169. Είμαι πεπισμένος ότι ένα διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα που εξασφαλίζει την διεθνή συνεργασία θα, είναι η πιο, θα κάνει πιο αποτελεσματικές τις δράσεις για την Βαλτική θάλασσα, για την αηφόρο ανάπτυξή της. Το bonus 169 ε, ε, εξασφαλίζει τη συμμετοχή 8 χρόνων. Υπάρχει όμως και μια άλλη χώρα, ε, συγκεκριμένα η Ρωσία, που μας ενδιαφέρει στα πλαίσια αυτού του ερευνητικού προγράμματος. Ε, το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να καταλήξει σε συγκεκριμένε προτάσει προ την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη τη Βαλτική θάλασσα και θα πρέπει να ασχοληθεί και με την μελλοντική ανάπτυξη μακροπεριφερειών που συζητήθηκε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να συζητήσουμε ανοιχτά και να. Ε, συγγνώμη, δεν ακούγεται πλέον ο μιλητής.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 Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω ότι η έρευνα στη Βαλτική θάλασσα θα πρέπει να ε, θεωρηθεί ένα στοιχείο συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εστιάζουμε την προσοχή μας σε διάφορες οριζόντιες ε, ε πτυχές ε, του θέματος που μπορεί να αφορούν και την Μεσόγειο, ε, παραδείγματος χάρη. υπάρχουν πολύ μεγάλες ε, εμπορικές δραστηριότητες που ε, σχετίζονται και με την Κίνα. Ελπίζω ότι η Βαλτική θάλασσα θα συνδεθεί ε, και με το Νότο μέσω του TNT και θα βρεθούν διάφορες δυνατές λύσεις. Ευχαριστώ η Επίτροπος για να απαντήσει εξ ονόματος της Κομισιόν για τις παρεμβάσεις αυτές. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Έκτην, η συγγήτρια και τα δέκα ε, μέλη που έλαβαν ε, το λόγο για να συζητήσουμε το θέμα. Είμαι ικανοποιημένη ότι ε, η πρωτοβουλία αυτή είναι στο 7 πρόγραμμα ε, και έχουν υιοθετηθεί. Είναι πολιτικό επίτευγμα για όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία bonus θα βοηθήσει τις χώρες της Βαλτικής να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τα περίπλοκα και κατεπήγοντα προβλήματα με συνέργειες και αποφεύγοντας την επικάλυψη των εθνικών προσπαθειών λόγω των πολιτικών γενικών προβλημάτων σε θέματα όπως η κλιματική αναγή, ενέργεια, πρέπει να συγκεντρωθούν οι πόροι και να υπάρξει συνεργασία. Το άρθρο 185, οι πρωτοβουλίες του παίζουν ρόλο σημαντικό για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Η πείρα που κερδίσαμε από τέτοιες πρωτοβουλίες θα μας επιτρέψουν να βρούμε καλύτερους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους συνεργασίας στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας καλύτερα τα προγράμματα. Όπως είπα, εδώ τον Ιανουάριο έχω δεσμευθεί για την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος έρμας, αλλά πρέπει να εργαστούμε μαζί μας σε ένα πνεύμα ενότητας και συνεργασίας για να έχουμε επιτυχία. Αυτό είναι ζωτική σημασία για την μελλοντική οικονομική ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να εξασφαλίσουμε ε, να γίνει σημαντικός ο πρωταγωνιστής στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχουμε την παρέμβαση της εισηγήτριας της κυρίας Έκα. Ευχαριστώ πολύ. Η πρωτοβουλία Bonus είναι ένα πρόγραμμα πιλωτικό βάση του άρθρου 185, όπως το είπατε και μπορώ να σας εγγυηθώ ότι όσοι συνεργαστούν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος που θα αισθανθούν τις συνέπειες άμεσα ή έμεσα, δεν θα αισθανθούν ότι δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούν αυτά τα ερευνητικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των διαφόρων χωρών μελών. Δεν είναι εύκολο, είναι μεγάλη πρόκληση, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει συντονισμός ανάμεσα στις διάφορες παραδόσεις στην έρευνα. 16 μεγαλειόμιλοι, 500 ερευνητές, 8 χώρες, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δει αν θα λειτουργήσει το σύστημα. Επιπλέον πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί σε αυτή την προσέγγιση. Θα χρειαστεί να δούμε αν οι απαιτήσει απέναντι στους ερευνητές και τα κράτη-μέλη είναι πολύ μεγάλες, θα πρέπει να ε, ληφθούν ε, πολιτικές ε, σκληρές, στεναρές και να υπάρξει μεγάλη πειθαρχία. Αλλά αυτά τα προγράμματα, τα ερευνητικά, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης αργότερα. Πρέπει σήμερα μαζί να αναλάβουμε αυτήν την ευθύνη για να επιλύσουμε τα προβλήματα της Βαλτικής και να αποτελέσουμε μοντέλο για άλλες περιοχές, για την Μεσόγειο επίσης ε, για τους πόρους γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα μοντέλο. Η Βαλτική θάλασσα αποτελεί μέρος της κουλτούρας μας, της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας. Από το τέλος της εποχής των παγετώνων σκεφτόμαστε τους Βίκινγκ, τους μεγάλους ταξιδευτές, σκεφτόμαστε και τον ψυχροπόλεμο. Είναι λοιπόν δική μας ευθύνη να διαχειριστούμε αυτήν την κληρονομιά. Ε, σκέφτομαι αυτές τις προκλήσεις, αυτά τα προβλήματα, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να σας ευχαριστήσω όλες και όλους. Η εργασία δεν έχει τελειώσει, ούτε καν όταν θα υιοθετηθεί αυτό το κείμενο και η υπογραφή. Τότε θα αρχίσει η εργασία ναι, μάλλον. Σας ευχαριστούμε κυρία Εκ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και η ψήφιση, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Περνάμε αμέσως στο ακόλουθο σημείο στην ημερησία διάταξη. Θέλω να σας επαναλάβω εδώ κάτι. Ότι